Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη της ε, συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, επαφείται σε μένα η άσκηση της Προεδρίας μια και ήμουν πρώτη αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Πάντως ο μοναδικός ε, σκοπός αυτής της ε, ολιγόλεπτης προεδρίας μου θα είναι η εκλογή του Προέδρου και τον, του Προέδρου της Επιτροπής μας. Ήθελα να ρωτήσω τις πολιτικές ομάδες ποιες είναι οι υποψηφιότητες που έχουν καταθέσει για το αξίωμα αυτό του Προέδρου της Υποεπιτροπής. Κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θα ήθελα να προτείνω ω πρόεδρο τον συνάδελφο Αγνό Ντονζόν. Μήπω άλλε πολιτικέ ομάδε έχουν δικό του υποψήφιο. Όχι. Οπότε μπορούμε να εκλέξουμε διαβοή στο συνάδελφο Αρνό Ντανζόν ω πρόεδρο της υποεπιτροπής μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την θέση αυτή και θα ήθελα να αποτίσω αφόρο τιμή στον κύριο Γκάου. Το γνωρίζετε όλοι, νομίζω ότι ήταν ε, αξιέπαινο το έργο του στην Προεδρία της Επιτροπής και μπορούμε να τον χειροκροτήσουμε θερμά. Θα προχωρήσουμε τώρα στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Pour la première vice-présidence, je demande θα ήθελα να μου προτείνουν οι πολιτικές ομάδες τον υποψήφιο ως πρώτο αντιπρόεδρο της Υποεπιτροπής. Merci, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εγκομιάσω τον πρώην πρόεδρο Φαβόγκαου για το αξιόλογο έργο του στην Προεδρία της Υποεπιτροπής. Και εκ μέρους ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Γιούστας Παλέτσκης. Λάθος, λάθος, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Monsieur, ε, Τον κύριο Κυριάκο Μαυρονικόλα για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου της Υποεπιτροπής. Συγγνώμη για το λάθος, τον κύριο Μαυρονικόλα. Μάλιστα, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για την πρώτη αντιπροεδρία της Υποεπιτροπής. Μπορούμε να εκλέξουμε διαβοή στον πρώτο αντιπρόεδρο ή ζητά κανείς μυστική ψηφοφορία. Όχι ο κύριος Μαυρονικόλας εξελέγει πρώτος αντιπρόεδρος υποεπιτροπής. Για τη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Ποια πολιτική ομάδα θα προτείνει αντιπρόεδρο. Ονομάζομαι Hans von και εκ μέρους των φιλελευθέρων θα ήθελα να προτείνω την κυρία Νόριτσα Νικολάη για τη θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου. Ε, είναι, βρίσκεται στην Αλοδαπή σε αποστολή, απουσιάζει. Ναι, όντω. Μα προειδοποίησε για την απουσία τη ε, κυρία Νικολάη. Υπάρχει άλλο υποψήφιο για τη θέση αυτή. Ή μήπω κανεί ζητά μυστική ψηφοφορία. Όχι, οπότε θα εκλέξουμε διαβοή στην κυρία Νικολάη. Για τον τρίτο αντιπρόεδρο, κυρία Γκόμες. Και τώρα θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Γιώργο Παλέτσκη εκ μέρου των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Θαυμάσια. Άλλε υποψηφιότητε δεν υπάρχουν, οπότε διαβοή εκλέγουμε και τον τρίτο μα αντιπρόεδρο, τον κύριο Παλέτσκη. Και τέλος θα εκλέξουμε τον τέταρτο αντιπρόεδρό μας. Oh, sorry. Ο κύριος Γκάλερ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προτείνω, δεν το βλέπω, είναι παρόν άραγε, το συνάδελφο Λίζεκ. Ζητώ συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Εκλέγουμε διαβοής και τον κύριο Λίσεκ ως τέταρτο αντιπρόεδρο της υποεπιτροπής μας. Après la constitution du bureau, nous allons faire un point sur le calendrier. Μετά τη συγκρότηση του Προεδρείου, θα εξετάσουμε το χρονοδιάγραμμα του δεύτερου εξαμήνου του 2009, που το έχετε λάβει. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα με αύριο το πρωί στις 9 και κατόπιν θα συνεδριάσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου μετά τις θερινές διακοπές. Η συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου ακυρώνεται. Γιατί εγώ θα είμαι στη Σουηδία και δεν μπορώ να παρήσαμε στη συνεδρίαση αυτή. Καλύτερα να την ακυρώσουμε από τώρα. Η συνεδρίαση 9ης Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, ακυρώνεται. Δεν έχουμε άλλα σημεία. Ραντεβού αύριο σε